ανάμεσα στις ε, θρησκευτικές ε, κοινότητες ε, και να συνοδεύσουμε τη χώρα στην οδό του πλήρους εκδημοκρατισμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουν κατατεθεί έξι προτάσεις ψηφίσματος. Τώρα θα περάσουμε στην ψηφοφορία. Ο συνάδελφος Μουνής έχει ζητήσει το λόγο της διαδικασίας. Παρακαλώ κυρία συνάδελφε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όσον αφορά το ψήφισμα για τη Ρωσία έχω να πω κάτι. Δεν νομίζω ότι θα είναι επίμαχη αλλαγή. Για την παράγραφο 18 να εφαρμόσει τι αποφάσει, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων Βορρική Ένωση να αντικατασταθεί αυτό. Αντί implement να λέμε adopt. Καλεί το Συμβούλιο να υιοθετήσει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελπίζω να μην υπάρχει πρόβλημα. Ja, aber wir haben keinen Paragraphen 18, oder? Nee, aber Μπλε κάρτα, κυρία Ογιουλέντ. επί της διαδικασίας. Δεν ξέρω, ίσως να μην κατάλαβα καλά από τη μετάφραση γιατί άκουγα τα ιστονικά. Δεν κατάλαβα πραγματικά τι έλεγε η συνάλφος. Μπορείτε να τα επαναλάβετε. Αν κατάλαβα καλά, κυρία Ογιουλαντ, θέλετε ε, κατάλαβα καλά, ήθελε η κυρία Συνάδελφο στο σημείο 18 να μπει ε, η λέξη adopt. Για, και θέλει να αντικατασταθεί η λέξη adopt ε, από τη λέξη να εφαρμόσει τι συμφωνίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν ξέρω, ίσως πρόκειται για ένα λάθος στο αγγλικό κείμενο μόνο. Κυρία Μονίθ, επαρκεί η λέξη εφαρμόσει για εσάς, σας επαρκεί. Ε, ναι, είναι η γερμανική εκδοχή, αν είναι σωστή στα αγγλικά. Η διαφορά είναι μεταξύ implement, σημαίνει να εκτελέσει κανείς να αντικατασταθεί από το adopt, υιοθετήσει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων αντί να εφαρμόσει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Περί αυτού πρόκειται. Ναι, αν κατάλαβα καλά, στα αγγλικά μιλάτε για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου τα οποία πρέπει να υιοθετηθούν και όχι να εφαρμοστούν. Adopted και όχι implemented. Υπάρχει κάποια αντίρρηση, δεν βλέπω καμία. Οπότε θα ψηφίσουμε με αυτή τη μορφή την παράγραφο 18. Ξεκινάμε την παράγραφο 8, αρχή, αρχικό κείμενο. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Παράγραφος 11 του αρχικού κειμένου σε τρία μέρη, μέρος πρώτο υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό μέρος τρίτο υπέρ. Ε, ρώτησα για το μέρος δεύτερο, λέει ο Όχι, μέρος τρίτο, υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Μετά παράγραφος 18 της κυρίας ε, Μονίτ, ε, όπως υποβλήθηκε υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Εκτιμώντας ΙΟΤ Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Το ψήφισμα στο σύνολό του υπέρ. Κατά. Αποχές. Ομόφωνα από ό,τι βλέπω. Να ακολουθεί η ψηφοφορία των έξι ψηφισμάτων για το Αζερβαϊτζάν για την περίπτωση Μαμάντοφ. Έχουμε το κοινό ψήφισμα 6 ε, ομάδων που θα αντικαταστήσει τα ψηφίσματα. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές δεκτό. Το ψήσιμο σύνολό του υπέρ κατά αποχές με μία ψήφο κατά. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία για έξι ψηφίσματα για το θέμα των Ροχίνγκια. Περνάμε πρώτα απ' όλα στο κοινό ψήφισμα που θα αντικαταστήσει τα 6. Παράγραφος 16 του αρχικού κειμένου υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Εκτιμώντας 16 τροπολογία είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Ψήφισμα σύνολό του όπως άλλαξε με ονομαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Παρακαλώ, ψήφισαν όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Με μία αποχή ομόφωνα δεκτό το ψήφισμα. Αγαπητοί συνάδελφοι, τα πρακτικά θα είναι στη διάθεσή σας στην αρχή της επόμενης ε, Συνόδου της Ολομέλειας. Ε, οπότε θα μεταβάσω στους αρμοδίους τα ψηφίσματα, δεν βλέπω καμία αντίρρηση και άρα διακόπτεται η συνοδού.